Καλώ ήρθατε στην συνεδρίαση τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, Δευτέρα βράδυ στο Στρασβούργο. Έχετε μπροστά την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει αίτημα για αλλαγή τη ημερήσια διάταξη. Βλέπετε ποιε γλώσσε έχουμε. Ελληνικά μπορούμε να μιλάμε και να ακούμε. Και επίση μεταδίδεται στο διαδικτύο. Να Καλώς ορίσω και την κυρία Βάλτερη, η οποία είναι καινούργια στη γραμματεία και είναι μάλιστα υπεύθυνη επικεφαλής της γραμματείας και θα μας ε, βοηθάει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Σας ξέρουμε και από την νομική υπηρεσία και επί σειρά ετών βοηθούσατε την Επιτροπή μας. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε στο σημείο 3 της ημερήσης διαταξής, την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Λεθνικού Συνεδρίου για την βοήθεια προς την Ουκρανία. Και στις 16 μέχρι 19 Μαΐου θα είναι η αντιπροσωπεία στην ε, Ουκρανία και θα σας ε, πω δύο λόγια γιατί ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Αν θέλετε λεπτομέρειες, έχετε μπροστά σας το έγγραφο. Να καλωσορίσω και τους εκπροσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Περιμέναμε λοιπόν την επεξεργασία των δύο εκθέσεων μέχρι ότου έχουμε και την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχουμε και τη Βάκεσαφ και τον κύριο Τσέλα από δική μα πλευρά, τον οποίο επίση καλωσορίζω. Ο κ. Φάσακα θα πάρει και παρά αυτά το λόγο για να μα παρουσιάσει την ειδική αυτή έκθεση. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξία κυρία αγαπητή είναι, αξιότιμη κυρία Γιώ, ε, αγαπητοί βουλευτέ, κύριε και κύριοι. Θα μιλήσω αγγλικά και γερμανικά. Αλλά η έκθεση είναι και συντεταγμένη στα αγγλικά, άρα προτιμώ τα αγγλικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι βρήκατε το χρόνο και μας δώσατε και την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε εδώ την έκθεση μας. Και πρωτού περάσω στις λεπτομέρειες της έκθεσης, θα ήθελα να σας συγχαρώ να σας συγχαρώ για το γεγονό ότι φτιάξατε ένα έγγραφο εργασίας στο οποίο βασίζεστε στα, στις δηλώσεις και στα πορίσματα και στις συστάσεις της δικής μας έκθεσης για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν. Νομίζω ότι αυτή είναι η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και Κοκομπού, ημών και ημών. Και έτσι βασίζεστε στην εργασία σα στη δική μα εμπειρογνωμοσύνη σα Δίνουμε λοιπόν τα απαραίτητα πορίσματα και τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να λάβετε πολιτικό πώ τι αποφάσει σα. Θα καταλάβετε ότι για μας, για τέτοια ευαίσθητα σημεία, δεν μπορούμε να απομακρυνόμαστε από τον πολιτικό κόσμο. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ειδική έκθεση από το 2016 για την ευρωπαϊκή αρρωγή προς την Ουκρανία, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερος που στην έκθεσή σας έχετε συμπεριλάβει ήδη τα πιο σημαντικά πολιτικά πορίσματα. Να ξεκινήσω τα, την παρουσίασή μας, την οποία και έχω παρουσιάσει, την έχω προετοιμάσει, συγγνώμη. Και καταρχάς θα ήθελα να σας πω ποια είναι η σημασία της έκθεσης αυτής. Όπως ξέρετε, η Ουκρανία είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, χώρες εταίρους, πολιτικός και οικονομικός, πως ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική αστάθεια, τα συνδέματα διακυβέρνηση, οι οικονομικά προβλήματα αποτελούν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της χώρας. Η ευρωπαϊκή οικονομική αρρωγή και αυτό ουσιαστικά πραγματευόμαστε σήμερα από το 2007 μέχρι το 2015 έφτασε τα 5 της ευρώ, 1,3 ευρώ σε επιδοτήσεις και 3,4 δις σε μακροοικονομικά δάνεια. Η ευρωπαϊκή αντίδραση λοιπόν στα όσα έγινε στο Μαϊντάν το 2014 ήταν η στιγμή που ξεκινήσαμε την έκθεση για την Ουκρανία. Μας ζητήθηκε. Είχαμε 11,2 δις ως πακέτο και βλέπετε ο συναδελφός μου έχει τα στοιχεία. Το θέμα του, από πλευρά του ελέγχου λοιπόν ήταν το εξή. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ήταν αποτελεσματική και αποδοτική στην αρρωγή που παρήχαν για τη μεταρρύθμιση και τη μεταμόρφωση του Ουκρανικού κράτους στον τομέα των δημοσιονομικών, και στην καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Οι δύο τομείς αυτοί θεωρήθηκαν οι δύο βασικοί τομείς για το μέλλον της ε, Ουκρανίας και στον τομέα της, ε, του αερίου που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το 2014 σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Και να ξεκινήσω με τα γενικότερα συμπεράσματα. Η ευρωπαϊκή αρρωγή προς την Ουκρανία ήταν εν μέρη αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την μεταμόρφωση της Ουκρανίας και του Ουκρανικού κράτους. Αλλά η ασταθής πολιτική κατάσταση, νομική κατάσταση και διοικητική κατάσταση περιορίσε την, το αντίκτυπο της ευρωπαϊκής αρρωγής. Από τα γεγονότα του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαστεί σε πιο συνεργατικό περιβάλλον, αλλά τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αρρωγής είναι ακόμα υποδιακύβευμα και η αντίδραση στην κρίση του 2014, η, η διάσωση του πακέτου των 11,2 δις ήταν μια λύση τις ανάγκης για να διατεθούν αυτά τα μεγάλα πόσα προκειμένου να βοηθηθεί η Ουκρανία και να αντιμετωπιστεί η καταπήγουσα οικονομική κατάσταση. Δεν υπήρχε προδιαγεγραμμένη στρατηγική εκείνη τη στιγμή εκείνη τη χρονική στιγμή. Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα και τα απορίσματα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δημοσιονομικών και την καταπολέμηση τη διαφθορά, η ευρωπαϊκή αρρωγή προ την Ουκρανία ήταν εν μέρη αποτελεσματική σε ό,τι αφορά δηλαδή την επίτευξη απτών και βιώσιμων αποτελεσμάτων στου δύο τομεί, αυτού που ανέφερα τα δημοσιονομικά και τη διαφθορά. Μέχρι το 2014 υπήρχε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα λόγω της ε, κυβέρνησης ε, και της σχετικής καθυστέρησης που υπήρχε και μετά από τα όσα έγιναν το 2014 παρόλα μάλλον τόσο συνέβησαν το 2014 τα, αποτελέσμα, αποτελέσματα είναι μάλλον μέτρια. Η αναστολή των δημοσιονομικών κονδυλίων και των μέτρων απελευθέρωσης ε, από το καθεστώς των θεωρήσεων ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τον τομέα του αερίου τώρα, η ευρωπαϊκή αρρωγή προ την Ουκρανία ήταν μερικώ αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη διακυβέρνηση του τομέα του αερίου και τη ε, εξασφάλιση του εφοδιασμού τη Ευρώπη. Μέχρι το 2014 η ευρωπαϊκή αρρωγή είχε περιορισμένο αντίκτυπο στην λειτουργία του τομέα του αερίου και είχε μεικτά αποτελέσματα. Ωστόσο, έχουν επιτευχθεί έκτοτε σημαντικά ορόσημα σε ό,τι αφορά μια σχετική νομοθεσία η οποία εγκρίθηκε τον Απριλίο 2014. Για παράδειγμα, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας χαρακτηρίζεται από δέσμευση το εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς και τις θέσεις που εκπροσωπούν σε ό,τι αφορά τη συλλογή σωστών δεδομένων, δεν υπήρχε σωστή παρουσίαση των δυσκολιών από πλευρά τη Ουκρανία. Και βάσει των πορισμάτων μα, έχουμε καταλήξει σε κάποιε πολύ σημαντικέ συστάσει. Η συστάση υπαριθμών 1. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ε, διαχείριση των δημοσιονομικών, στον διάλογο και στη διαδικασία διαλόγου με την Ουκρανία να υπάρχει και ένας ενισχυμένος διάλογος για θέματα τέτοια διαχείρισης των δημοσιονομικών, προκειμένου να υπάρχει σωστή στρατηγική και να εφαρμοστεί αυτή το συντομότερο δυνατό. Δεύτερη σύσταση. Βελτίωση του σχεδιασμού των συνθήκων σε ό,τι αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας. Οι δείκτες για την ε, δημοσιονομική υποστήριξη θα πρέπει να ορίζονται βάσει των σωστών όρων και θα πρέπει οι μελλοντικοί στόχοι να είναι σε συνεργασία με τους στόχους συνολικά. Και θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της μόχλευσης παιδοπολιτικής και της ανάγκης να υπάρχει γρήγορη παροχή αρρωγής. Τρίτη σύσταση σε αφορά την ίσχυση της παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αρρωγής που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Να υπάρχει εναρμόνιση της ε, προσέγγιση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα προγράμματα παροχής ε, δημοσιονομικής αρρωγής. Τρίτη, τέταρτη μάλλον σύσταση, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή και βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Να υπάρχει αρεσιμότητα. Να δίδεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο να υπάρχει σωστή εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων και να ε, εκτιμούνται και να αξιολογούνται αυστηρά οι όροι για την ε, χορήγηση των, ε, α, της αρρωγής. Πέμπτη σύσταση σε ό,τι αφορά τον τομέα του αερίου. Να ληφθούν βήματα προκειμένου η ευρωπαϊκή αρρωγή στην Ουκρανία να είναι πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τον τομέα του αερίου. Να υπάρχει καλύτερη ανάλυση και επαληθεύση των δεδομένων να είναι πιο ακριβή η πληροφορία ακόμα και υπό δεσμενείς συνθήκες. Αυτά θέλαμε να σας παρουσιάσουμε αναφορικά με την έκθεσή μας, η οποία καλύφθηκε από τη δημοσιότητα και από τον τύπο και ε, συγκεντρώσε μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πούμε, από τον τύπο. Δεν είναι θέμα και δεν είναι στο πεδίο της εντολής μας να ασχολούμαστε με τον τύπο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι υπήρξε μεγάλη παρερμηνία από πλευρά των μέσων δημοσιότητας, γιατί ουσιαστικά το μήνυμα ήταν προς ε, το κοινό ότι η έκθεση μας έλεγε ότι η Ουκρανία είναι η πιο δεθαρμένη χώρα. Δεν είναι όμως το πεδίο εφαρμογή μας, στο πεδίο εφαρμογής του Ελεκτικού συνεδρίου να σχολιάσουμε τη διαφθορά μιας χώρας. Απλά επισημάναμε ότι βάσει των ε, διεθνών δεδομένων θα έπρεπε να γίνει μια σχετική ανάλυση. Αλλά αυτά τα στοιχεία που σας είπα δεν ήταν δικά μας, ήταν στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας, Transparency International, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα διαφθοράς. Είχαμε την αίσθηση όμως ότι οι δύο βασικοί τομείς ήταν η διαχείριση των δημοσιονομικών και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτοί οι δύο τομείς θεωρήσαμε ότι ήταν οι τομείς προτεραιότητας για τη χώρα, προκειμένου η χώρα να μετατραπεί σε μια χώρα δυτική, δυτικοευρωπαϊκή, σε ό,τι αφορά θέματα διακυβέρνησης και οικονομίας. Αυτά και ευχαριστώ, Πρόεδρε. I'm looking forward to... Και προσβλέπω φυσικά στις ερωτήσεις σας και στα σχόλιά σας για την έκθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγητής κύριος Τσέλερ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε επίσης πολύ τον συνάδελφο κύριο Φάτσακας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους συνεργάτες του για αυτή την έκθεση σε μια πολιτικά πολύπλοκη διαδικασία, δηλαδή την ενίσχυση που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία και συνεχίζει να παρέχει ε, σε μια πολιτικά δύσκολη συγκαιρία. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδριού περικλεί το χρονικό διάστημα από 2007 έως 2015 ε, δηλαδή την παλιά περίοδο μέχρι το 2013 αλλά την ε, υπερβαίνει ε, εξετάζοντας και τα δύο τελευταία χρόνια μέχρι το 2015. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία μέχρι το 2013 διαπιστώνουμε και αυτή είναι και εξακρίβωση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι οι βοήθειες που δόθηκαν στην Ουκρανία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, δηλαδή το 1994, δόθηκαν οι βοήθειες αυτές, αλλά συχνά ήταν δύσκολο να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα ε, της ε, βοήθειας αυτής ε, στο πλαίσιο αυτής της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. η συμφωνία αυτή ε, ε, ε, έμελε να αντικατασταθεί από μια συμφωνία εταιρική σχέσης και στη συνέχεια υπό την προεδρία του κυρίου Γιαννουκόβιτς η συμφωνία αυτή σύνδεσης της Ουκρανίας και κατόπιν της πίεσης της Ρωσίας δεν μπόρεσε να υπογραφεί. Ε, και αυτό οδήγησε σε ένα μαζικό κίνημα στην Ουκρανία το οποίο έγραψε ιστορία με το Μαϊντάν κλπ όταν ε, οι πολίτες της Ουκρανίας δεν ήθελαν να αποδεκτούν ο δρόμος ε, προσέγγισης της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συνεχίσει. Γιατί βεβαίως η Συμφωνία Σύνδεσης της Ουκρανίας θα ήταν ένα περαιτέρω ορόσημο στην προσέγγιση της, ε, στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας. Ε, υπήρξαν ε, πολλά θύματα μεταξύ των πολιτών και η εξέγερση αυτή σημείωσε μια υποτυχία γιατί υπήρξε μια πολιτική αλλαγή στην Ουκρανία και η νέα κυβέρνηση και ο ενεκλεγής πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία σύνδεσης ε, κάτι που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την θετική υποχρέωση παροχής περαιτέρω βοήθειας ε, στην Ουκρανία 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για, ξεκινώντας από το 2014 και για 11 χρόνια. Στη συνέχεια Ε, υπήρξαν άλλες ε, πολιτικές ε, αλλαγές, αλλαγές στην ηγεσία της Ουκρανίας και είδαμε ότι τελικά οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν και πολύ σημαντικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες τελικά δεν εφαρμόστηκαν με την αναγκαία προσοχή, η συστηματικότητα. Κάτι που επίσης το επισημαίνει το ελεγκτικό συνέδριο ε, και το οποίο εξέτασε προσεκτικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον τομέα του φυσικού αερίου, όπου η Ουκρανία ήταν άμεσα εξαρτημένη από, τον, ε, από τη Ρωσία στον αφορά τον εφοδιασμό φυσικό αέριο και συνεχώς υπήρξε μια διάνεξη όσον αφορά τις πληρωμές του φυσικού αερίου από τη μία πλευρά και από την άλλη το γεγονός ότι ο τομέας του αερίου στην ε, Ουκρανία αποτέλεσε μία πύλη για ένα παράθυρο για διαφθορά και εκ μέρους ε, ολιγαρχών της Ουκρανίας οι οποίοι ε, προσπάθησαν να μοιράσουν την λία στην Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά τους ε, ευρωπαϊκούς αγωγούς, έχουμε πλέον μια σχετική εποπτεία για το τι γίνεται, έναν έλεγχο και υπήρξε μια σταθεροποίηση του εφοδιασμού του αερίου ε, στην Ουκρανία, με αέριο στην Ουκρανία. Αλλά τώρα διολυσταίνει η χώρα σε μια άλλη σύγκρουση μετά την αντισυνταγματική προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, αποσχιστικά κινήματα στο Ντονέτσκ, στην Ανατολική περιοχή, ε, που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και όλα αυτά όθησαν τη χώρα στα πρόθυρα μιας εμφύλιας σύραξης και στις χώρες αυτές ε, τελικά ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος ο οποίος ε, επίσης οδήγησε σε πολλούς ε, νεκρούς και στην ε, αφέμαξη των πόρων της χώρας. Θα πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ούτως ώστε να σταθεροποιήσει τις δομές της και να μπορέσει να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις και να μπορέσει να προσμετρήσει την πρόοδό της τους ευρωπαϊκούς γνώμονες. Αλλά από την άλλη, βεβαίω, ε, ε, θα πρέπει να ασκήσουμε μια κριτική στην Ουκρανία όσον αφορά την ε, καθυστέρηση όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων, γιατί οι ενισχύσεις έχουν ακριβώς σαν στόχο να οδηγηθεί η Ουκρανία προς τον εκδημοκρατισμό και τον εξυγχρονισμό. Ε, γι' αυτό ε, λυπόμαστε ότι, ε, για το γεγονός ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες αμφίστανται ακριβώ στον εκδημοκρατισμό και τον εξυγχρονισμό της χώρας. Χαιρετίζουμε τις, τις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, αλλά έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να συνδεθούν τα χρήματα αυτά με την προσπάθεια εκ μέρους της Ουκρανικής κυβέρνησης να βελτιώσει την ε, κατάσταση των εσόδων στη χώρα και την ε, δημιουργία ε, κάποιων διαφανών δομών, φορολόγηση για παράδειγμα, η οποία μπορεί να προσεγγίσει και τους ολιγάρχες. Να τους υποχρώσει δηλαδή να πληρώσουν και να φορολογηθούν και εκείνοι. Ε, υπάρχουν ε, ε, πάρα, πολλοί οργανισμοί οι οποίοι συστάθηκαν με την Ευρωπαϊκή Συνδρομή και οι οποίοι έχουν σαν στόχο να καταπολεμήσουν την διαφθορά και οι οποίες έχουν προσωπικό το οποίο διορίζεται από την Ουκρανική κυβέρνηση και χρηματοδοτείται και από την Ουκρανική κυβέρνηση, κάτι το οποίο δημιουργεί βεβαίως κάποιες αμφιβολίες. Χαιρετίζουμε το ότι όπως είπε και η Πρόεδρος, ε, το περασμένο έτος είχαμε μια αποστολή με την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμού στην Ουκρανία και εκεί μας ανέφεραν ότι δύο τρίτα των ε, δικαστών στην Ουκρανία είναι εκατομμυριούχοι. Ε, και των νομικών παραστατών. Και άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να γίνουν ε, πάρα πολλά πράγματα ώστε να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και να μπορέσουν οι πολίτες ε, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη προς το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Επίσης το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να ελέγχεται πιο συστηματικά ώστε να μειωθούν και οι ροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό που συνεπάγονται ε, μια ε, χρεοκοπία τελικά του τραπεζικού συστήματος και ε, Ελπίζουμε η, μακροχρηματοδοτικές, η μακροχρηματοδοτική συνδρομή, η οποία έχει χορηγηθεί και στο παρελθόν, να συνεχίσει να δίδεται στην Ουκρανία και αυτή η συνδρομή δόθηκε στο παρελθόν, ώστε να προστατευτεί το σύστημα της ε, Ουκρανίας από την ε, κατάρρευση. Έχει 20% πληθωρισμό, ήδη είναι ψηλό, αλλά θα μπορούσε να είναι, όπως ήταν και στο παρελθόν, 150%. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, κάτι το οποίο δεν ήταν ορατό μέχρι στιγμής ε, στο παρελθόν. Και επίσης απαιτούμε η χορήγηση της ε, οικονομικής ε, βοήθειας να συναρτάται έτσι όπως ε, αναφέρει και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου να συνδεθεί με μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας αυτής της βοήθειας και βεβαίως ε, ε, αυτό το οποίο χρωστάει η Ουκρανική κυβέρνηση είναι και μία αποκέντρωση της ε, διοίκησης της χώρας. δεν υπάρχουν ικανές ε, σταθερές διοικητικές δομές στο επίπεδο των περιφερειών όπως για παράδειγμα η περιοχή του Λέμπερκ ή το ίδιο το Λέμπερκ έχουν ε, εξελιχθεί ε, θετικά και υπάρχουν εκεί κάποιες αποκεντρωμένες δομές και ίσως οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν ε, μοντέλο για άλλες ουκρανικές ε, περιφέρειες και να τους παράσχουν ενδεχομένως και τεχνική συνδρομή και στήριξη. Ε, αυτά μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την σχέση με την Ουκρανία και κυρίως να έχει θετικά αποτελέσματα για τους ε, πολίτες της χώρας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη ε, επισκόπηση για το ταξίδι πέρσι το Μάιο στην Ουκρανία, γιατί από τη μία θα πρέπει ε, σε δέκα λεπτά να κάνω την ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και θα ήθελα να σας πω ότι βρήκα εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι σε αυτή την αποστολή των 7 ήταν, μόνο τρία τελικά τα μέλη, ενώ αρχικά είχαν, είχε προγραμματιστεί μια αποστολή 7 μελών. Ε, δηλαδή είμαστε πολύ λίγοι τελικά ε, και τόσο λίγοι που δεν ήταν δυνατόν να στεφθεί με επιτυχία η αποστολή αυτή γιατί έπρεπε να σχηματίσουμε μια σωστή αίσθηση για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη χώρα και θεωρώ ότι είναι σημαντικό και η Ουκρανία πραγματικά αξίζει της ε, δικής μας ε, βοήθειας και ε, εν ώψη των τεράστιων ποσών που δίνουμε στη χώρα αυτή είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή αίσθηση για το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή. Χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριο Βάγνερ από την DG και άλλοι συνάδελφοι μας πούν ε, κάποια πράγματα για την ε, χρήση των ε, κονδυλίων. Ξεκινήσαμε από το Λέμπερκ, ωραία είναι εκεί, αλλά υπάρχουν και άλλες σημαντικές περιοχές που ίσως είναι πιο χαρακτηριστικές για την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στην Ουκρανία. Βεβαίως ήταν θετικό να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που λειτουργούν σωστά. Πήγαμε και στο Κίεβο και είχαμε και εκεί μια εμπειρία και ίσως ε, μπορούν, είναι δυνατόν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις για το γεγονός ότι αυτή οι αόρατοι ε, ολιγάρχες τελικά ε, εμφανίστηκαν αλλά για να μας πούν πράγματα τα οποία ήθελαν να ακουστούν. Ε, δεν ξεχάσαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο ότι πρόκειται για μια χώρα που βρίσκεται στον πόλεμο ε, και βεβαίως υπάρχουν τεράστιες ε, ανάγκες οι οποίες είναι μετρήσιμες ε, κάθε μέρα όσον αφορά την καταβολή των συντάξεων, ε, την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν κάτω από εντελώς αναξιοπρεπείς συνθήκες και παλεύουν για να πάρουν τη συντάξη τους και προσπαθήσαμε και εμείς να δείξουμε κάποια κατανόηση από την πλευρά μας και θα ήθελα πάρα πολύ να επαναληφθεί αυτό το ταξίδι γιατί θα ήταν πολύ σημαντικό εκεί να έχουμε πραγματικά, να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιες γνώσεις και μια αίσθηση για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Είδαμε ότι οι Πολωνοί φίλοι έχουν πολύ στενές σχέσεις με την Ουκρανία και υπάρχει και διασυνοριακά κάποιες ε, ε, υπάρχει κάποια κίνηση η οποία ακριβώς στο επίπεδο αυτής της σχέσης γειτονίας έχει θετικά αποτελέσματα. Ε, έχουμε από τη μία είχαμε μία, δύο όψεις ε, μιας εμπειρίας πραγματικά φρικιαστικές εμπειρίες όσον αφορά την τεράστια αντίσταση σε αλλαγές στην Ουκρανία όπου όλα γίνονται μόνο εφόσον ασκηθεί τρομακτική πίεση. Υπάρχουν βεβαίως μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, αλλά η αντίσταση είναι πιο ισχυρή από τη βούληση των μεταρρυθμίσεων. Και από την άλλη είδαμε ότι η συνεχής πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλα αυτά είχε θετικά αποτελέσματα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Γραμματεία γιατί πραγματικά ήταν ενδιαφέρον το ταξίδι και θα ήθελα, και θα ήθελα να επαναληφθεί αλλά να γίνει με 7 μέλη, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν ε, σημαντικό να ενισχύσουμε την ε, παρουσία μας εκεί. Ο κύριος Βαλέσα θέλει πρώτος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο εισηγητής για την ίντα όσον αφορά την Ουκρανία και έχω δύο τίνα που έχω να σας αναφέρω που είναι σημαντικά. Ένας από τους βασικούς τομείς που καλύπτουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και επίσης προβλέπονται ε, κάποιες ειδικέ διοκτικές αρχές όσον αφορά το να θεσπιστούν αυτά τα εγκλήματα και επίσης να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αποσπάσουμε κάποια τα αποτελέσματα με αυτά τα μέτρα τα οποία να πιάσουν τόπο. Εσείς τι θα συνιστούσατε όσον αφορά την διαφθορά, τι θα προτείνατε. Ας πούμε να έχουμε κάποια αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων από το αντίστοιχο σύστημα όσον αφορά ε, κάποια στοιχεία για δημόσια περιουσία. Τώρα επίσης τι γίνεται όσον αφορά την ε, εκταμίευση της μακροοικονομικής ενίσχυσης και ε, εννοώ το να υπάρξει κάποια ρύθμιση, κάποια νομοθεσία για την ενέργεια. Δεν έγινε αυτό από το Κοινοβούλιο. Αλλά έχουμε επίσης και την απαγόρευση εξαγωγής ανεπεξέργαστης ξυλίας. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ιδίως όσον αφορά αυτήν την απαγόρευση για την ξυλία είναι κατά του ΠΟΕ και οποιασδήποτε εμπορική συμφωνίας ε, γιατί πάμε για κάποιο είδους ασύμετρες εκχωρήσεις. Θα πρέπει επομένως αυτοί οι φραγμοί στο εμπόριο να αρθούν κατά τον οικονομικό έλεγχο. Εσείς τι είδους φραγμούς εντοπίσατε. Σας ευχαριστώ κύριε Κινίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου και μπράβο για την έκθεσή του επίσης και τον κύριο Τσάιλ γιατί εις βάθος και ολοκληρωμένα εργάστηκε νομίζω ότι αυτή η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ ακριβής είναι τεκμηριωμένη όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο πλευράς βοηθείας. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα υπάρχοντα προβλήματα. Θα πρέπει να τα επιλύσουμε με ένα πρόγραμμα αρρωγής που να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό και έτσι να βοηθήσουμε στην οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας. Όπως έχει διαπιστωθεί υπάρχει αργή πρόοδος. Είχαμε βέβαια την ε, μεγάλη αλλαγή του 2014. Και σαν πολλές δυσκολίες οι μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και την ε, κατανόηση της διαφθοράς. Αλλά έχουμε και προβλήματα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει 100% αλλά νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικά τα όσα έχουν γίνει. Μια που είναι οι καταστάσεις δύσκολες, είναι κατάσταση επίγουσας ανάγκης, κυρίως μετά τα γεγονότα του 2014. Άρα χρειάζεται αποτελεσματική και ξεκάθαρη στρατηγική με βάση την αιρεσιμότητα και τους σχετικούς κανόνες. Να είμαστε ρεαλιστές, να έχουμε υπόψη το πόσο ευάλωτα είναι τα αποτελέσματα. Άρα, γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε τη χώρα σε αυτή τη διαδρομή ανάπτυξης. Η πολιτική συγκυρία παραμένει περίπλοκη, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα πιάσουν τόπο, θα ριζώσουν οι αλλαγές που ήδη έγιναν. Νομίζω ότι η αξιολόγηση του ελληνικού συνεδρίου είναι πολύτιμη για την Επιτροπή. Θα ήθελα να πω από τη συνέχεια τον όσων είπε ο προλαλή σα ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την ερεσιμότητα σε σχέση με την χρηματοδότηση για την μαρκοοικονομική αραγή. Όσον αφορά την δεύτερη δόση των ενισχύσεων που προβλέπετε. Περισσότερες λεπτομέρειες επομένως. Τι προϋποθέσεις προβλέπονται, τι απαιτείται για να δοθεί αυτή η δεύτερη δόση. Uh, thank you for that. We seem to be merging uh, items 3 and items 4. Από ό,τι φαίνεται συζητούμε ταυτόχρονα το 3 και το 4. Έχουμε αυτή την ειδική έκθεση όσον αφορά την ε, Επιτροπή στην Ουκρανία. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό αυτό. Οπότε τώρα μπορείτε αντίστοιχα να μας πείτε τι γίνεται για το θέμα, τι έγινε στην ε, αποστολή. πολύ έχουν στο λόγο μεταξύ των οποίων η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω το Ελληνικό Συνέδριο για αυτήν την ε, σημαντική έκθεση. Ήδη αναφέρθηκε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Κυρίως ο κύριος Τσέλερ μας τα ανέλησε και εγώ έχω παρακολουθήσει τι γίνεται ιδίω όσον αφορά τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη γιατί εργάζομαι στα πλαίσια της ε, ε, του γραφτού φορέα Euronest. τι μόχλευση τα διεθνή θεσμικά θα μπορούσαν να ασκήσουν τόσο ώστε να υπάρξουν προς το καλό κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Τράπεζα Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήδη έχουν ε, θετική εμπειρία. Ιδίως αφορά τη μεταρρύθμιση για το φυσικό αέριο, που εκεί υπάρχουν ε, διάφανες συνθήκες στις κρατικές προμήθειες και τέτοια θέλουμε. Τέτοιου είδους κοινή μόχλευση, κάτι άλλο. Κατά πολέμηση της διαφθοράς στο υψηλό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Σχετίζεται δε με αυτόν τον έκτακτο διαρισμό και τον πρόεδρο Προσέγκο την Άνοιξη. Διόρισε ένα νέο γενικό εισαγγελέα που ήταν πολιτικός. Και ο κ. Λουτσέγκο είχε κάθε ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι μερόληπτος, αλλά δεν ισχύει ακριβώς κάτι τέτοιο. επομένω. θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς. Θα ήθελα δύο λόγια όσον αφορά το τι προοπτικές έχει το θέμα. Τέλος. Η ηλεκτρονική δήλωση ήταν τόσο αποτελεσματική που πάρα πολλοί εκατοντάδες δικαστών αποφάσισαν να πάνε σε πρόορη σύνταξη αντί υπογράψουν αυτή την δήλωση. Νομίζω και άλλες χώρες μπορούν να αντιλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα. Να, μια σωστή αφετηρία για την κάθαρση, α πούμε αυτή τη σκληρή λέξη, για την κάθαρση ευμένως, στην δικαιοσύνη. Όλα αυτά μας είπε ο κύριος ε, Τσέλερς στις συστάσει του Πάντω, Νομίζω ότι καλά τα λέει το Ελληνικό Συνέδριο και θα πρέπει να υπάρχει αυτό το είδου η κοινή μόχλευση. Και δούμε τι θα γίνει επίση και με την υπηρεσία του Γενικού Εισαγγελέα. Ευχαριστώ, λέει ο Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, είναι ενδιαφέρον που βρισκόμαστε εδώ. Είμαι η πρώτη συνεδρίαση ω πλήρε μέλο τη Επιτροπή και αντικαθιστώ τον κύριο Τόιρερ. Δεν είναι φυσικά εύκολο Πώ να γεμίσω τα παπούτσια του, όπως λέγει η φιλανδική παροιμία. Θα κάνω τι μπορώ. Να πω και δύο λόγια για την ε, ειδική αυτή έκθεση. Να ευχαριστήσω το μέλος του Αλεκτικού Συνεδρίου του Κρυφά που ήταν πρώην μέλος εδώ. Και είστε και καλός παίκτης του τέννις. Παίζετε και καλό τέννις. Σας ευχαριστώ όμως τώρα για την ισορροπημένη αυτή και καλή έκθεση που μας βοηθάει να καταλάβουμε πώ θα βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή αρρωγή προ την Ουκρανία στο μέλλον. Και τον κύριο Γιώργη Μιτσέλερ να ευχαριστήσω για την καλή συμβολή του που μα βοηθά για τη δουλειά μα στην Επιτροπή. Καταρχά, η Ουκρανία έχει περάσει δύσκολε περιόδου. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Σε ό,τι αφορά την πορτοκαλί επανάσταση σε ό,τι αφορά την, ε, το θέμα με την, ε, τα σύνορα της με τη Ρωσία και να μην ξεχάσουμε και το 2008 την οικονομική κρίση της Ουκρανίας. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για μεταρρυθμίσεις, η Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί την πιο δεθραμένη χώρα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία και για να καθοδηγήσει και για να επιλύσει τα προβλήματα της με τη Ρωσία. Να τονίσω την διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα της ευρωπαϊκής αρρωγής προς την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ορατό και θα πρέπει η παρακολούθηση των εφαρμογών αυτών, της εφαρμογής αυτής των μέτρων, να είναι πιο εντατική για να υπάρχει πρόληψη της διαφθοράς σε όλες τις μορφές. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι συχνά εξίσου αποτελεσματικό όπως και τα χρηματοοικονομικά κίνητρα. Και είμαι πεπισμένος ότι μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τη δημόσια διαχείριση. Ευχαριστώ. Και έχω μπει και εγώ στο κατάλογο για να μιλήσω. Γιατί πήγα στην αντιπροσωπεία στην Ουκρανία πέρσι το Μάιο. Έχει περάσει καιρό. Και προσπαθώ να θυμηθώ τα τι συζητήσαμε τότε. Και τι με εντυπωσίασε. Κάτι που το οποίο συζητήσαμε ήταν η διαφθορά και το πλαίσιο κατά τη διαφθορά στο οποίο εφαρμόζεται τώρα συναντηθήκαμε με διάφορα σώματα κατά της διαφθορά και μικιό. Και αυτό αφενός μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην κουλτούρα της Ουκρανίας, αλλά αντιθέτως ακούσαμε και πάρα πολλά για την διαφθορά. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ερώτημα προς τον κύριο Βάγνερ κατά πόσον έχει την αίσθηση ότι έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση ή κατά πόσον συνεχίζουν τα πράγματα στο ίδιο επίπεδο. Το δεύτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δίδονται προς την κεντρική κυβέρνηση. Φυσικά είναι δύσκολο να ανοιχνευτούν αυτοί οι πόροι. Και το θέσαμε αυτό σε ερώτημα στην επίσκεψή μας η απάντηση που λάβαμε είναι μάλλον καλή. Ότι ξέρετε έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ουκρανία. Δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα παρακολουθούμε κάθε ευρώ στην Ουκρανία. Δεν μπορείτε να μας ζητάτε κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν το θέμα είναι κατά πόσο επιμείνουμε επιμένουμε στο θέμα αυτό ή κατά πόσο να αποδεχόμαστε την εξήγηση ότι η Ουκρανία στην παρούσα φάση δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να δώσει πιο πολλά στοιχεία. Και να δώσω το λόγο στην κύριο Βάγνερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνδεθήκαμε και στην Ουκρανία και ίσως να έχει κάποιε απαντήσει για τα θέματα που θέσαμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που σχολίασε την έκθεση του ελέγχου. Το πιο βατικό στοιχείο είναι, όπως είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δεχτεί όλες τις συστάσεις της έκθεσης. Αυτό καταδεικνύει ότι για πολλά ζητήματα που περιλαμβάνονται στο, στην έκθεση υπάρχει ευρεία συνένεση. Ας πάμε και ένα βήμα πίσω όμως και να τονίσουμε και πάλι την πολιτική σημασία των ζητημάτων αυτών σε ό,τι αφορά την παροχή αρρωγή στην Ουκρανία. Υπήρχαν πολιτικέ εξελίξεις, όπως είπε ο εισηγητή, ελήφθησαν πολιτικές αποφάσεις για να υποστηριχθεί, να σταθεροποιηθεί και να βοηθηθεί η χώρα. Και εδώ υπησέρχονται οι ευρωπαϊκοί φορείς ό,τι αφορά την εφαρμογή όλων αυτών. Και κατανοούμε ότι αυτό αναγνωρίζεται στην έκθεση της αποστολής καθώς και στην έκθεση του ελέγχου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπογραμμίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις όλες τις αλλαγές που έχουν ήδη λάβει χώρα από την ε, επανάσταση του Μαϊντάν. Να μην ξεχνάμε ότι από πλευρά σε πρόκειται για μια χώρα η οποία ήταν στο χείλο ε, τη καταστροφή οικονομικά. Ο κόσμο πέθανε. Και τότε η κυβέρνηση ξεκίνησε σχετικά άμεσα τις μεταρρυθμίσεις που δεν είχε γνωρίσει η χώρα την προηγούμενη 20η-30η ετία. Να το θυμόμαστε αυτό, ότι επί σειρά δεκαετιών η Ουκρανία ήταν μέρο του Σοβιετικού κράτους. Και έχασαν δεκαετίε ολόκληρες μετά την εξαρτησία. Μόνο από το 2014-2015 έχουν ξεκινήσει οι μεταρρυθμίσεις. Το αναγνωρίζουμε λοιπόν αυτό και αναγνωρίζουμε και τα όσα λέει το δικαστήριο, ότι πρόκειται για μια καταπήγουσα κατάσταση, κατάσταση έκτατης ανάγκη. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει οι καταπήγουσες καταστάσει απαιτούν και καταπήγοντα μέτρα. Και μόνο στη συνέχεια μπορούμε να ακολουθήσουμε πιο στρατηγικές λύσεις. Άρα αναγνωρίζουμε το τι συνέβη, το τι έχει ήδη επιτευχθεί και θα δώσουμε και μερικές απαντήσεις στο τέλος. Και ύστερα να δούμε τι έχει γίνει μετά την πρώτη φάση της αθροποίησης. Και αυτό γιατί. Γιατί πρωτού δημοσιευτεί η έκθεση, οι τελευταίες 20 μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε μια έκθεση που επικεντρώθηκε στα θέματα διαφανούς και υπεύθυνης διακυβέρνησης και τι περιλαμβάνει. Αποκέντρωση. Σημαντικό για το μέλλον της χώρας, προκειμένου να λάβουν ε, αξία και εξουσία οι δήμοι οι κοινότητες, οι περιφέρειες και εδώ βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει σωστή εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατά της ευθοράς, ένα νέο πρόγραμμα συστάθηκε, το οποίο ξεκινάει να εφαρμόζεται τις ημέρες αυτές που συστάθηκε από δανέζικέ υπηρεσίε, από διεθνεί εμπειρογνώμονε και επικεντρώνεται ακριβώς στου τομείς του οποίους αναφέρατε. Δηλαδή, οικοδόμηση θεσμικών των θεσμών, αλλά και θεσμική διαμόρφωση των, των νέων αυτών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πλέον νέες υπηρεσίε οι οποίε θα λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα. Ύστερα, έχουμε και αντίστοιχα προγράμματα για το κρατό δικαίου. Κάτι άλλο που δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν οι οικονομικές απόψεις ε, και οι οικονομικές προοπτικές της χώρας. Στην Επιτροπή είμαστε πεπισμένοι ότι αν η δεύτερα τα δικαστικά συντήματα τα θέματα κρατός δικαίου ρυθμιστούν, θα ακολουθήσει και η οικονομική κατάσταση, γιατί όπως σας είπατε υπάρχουν πολλά λεφτά στη χώρα, και εκτός χώρας δηλαδή, που θα σταθεροποιούσαν την κατάσταση και ο πληθωρισμός για παράδειγμα είναι στο 10-10% και όλοι αυτοί οι φορείς θα επέστρεφαν στη χώρα. Σε ό,τι φορά τη μεταρρύθμιση επίσης ε, του δημοσίου τομέα. Αναφέρθηκε και ο εισηγητής και η κυρία Γκρέσλε στο θέμα αυτό για την, ε, να υπάρξει νέο αίμα στην Ουκρανία στο σύστημα. Όλα αυτά λοιπόν τα παρακολουθούμε ενεργά. Και οι εργασίες αυτές βρίσκονται υπό εξέλιξη. Όπως είπα και προηγουμένως, συμφωνούμε με τις συστάσεις. Υπάρχουν και σχέδια δράσεις τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Και θα ακολουθήσουν και άλλες συστάσεις. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάνα δυο από τι ερωτήσει που θέσατε. Και μετά θα μπορούσε να πάρει το λόγο και ο συνάδελφο για να συνεχίσει. Σε ό,τι αφορά τι διεθνεί οργανώσει και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διεθνεί οργανώσει και το καθεξή. Από ό,τι ακούω, δεν είναι πολλέ οι χώρε με τι οποίε είναι τόσο στενή η συνεργασία. Είναι διαφορετική η κύκλη, ασφαλώ και τα νομικά συστήματα, αλλά εργαζόμαστε ε, στενά σε ό,τι αφορά την ΕΤΕΠ, την ΕΚΤ, το ΔΝΤΟΥ και η νέα στρατηγική, για παράδειγμα, για τη διαχείριση της δημοσιονομικών. Αυτό παρακολουθήθηκε και από την ε, Παγκόσμια Τράπεζα και από τους α, ε, άλλους παγκόσμιους δωρητές. Υπάρχουν ε, πολλά συντονισμένα προγράμματα λοιπόν και με, τα, με τις για παράδειγμα που μας επιτρέπουν να διπλασιάζουμε την χρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά το αέριο, σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο και την καταπολέμηση τη διαφθορά. Και εκεί συνεργαζόμαστε στενά. Να πούμε δύο λόγια για την κοινωνία των πολιτών, που αποτελεί και ένα από του βασικού φορεί που προωθούν τι ε, μεταρρυθμίσει στην χώρα. Γιατί υπάρχουν και οι παλαιότεροι, οι οποίοι προωθούν το παλαιό σύστημα, αλλά παράλληλα έχουμε και πίεση από εξωτερικούς παράγοντες στην Ουκρανία και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να παραμείνουν στο σωστό δρόμο οι κυβερνήσεις. Τώρα, κάποιοι τομείς όπου πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές να σας αναφέρουμε. Ο τραπεζικός κλάδος αναφέρθηκε. Εξακολουθεί να αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση αν δούμε όμως το τι έχει συμβαίνει, τι έχει ήδη συμβεί σε ό,τι αφορά τράπεζες ε, που ουσιαστικά καταχρούνταν το δημόσιο χρήμα, έχει συμβεί, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Αυτό υποτιμάται ενδεχομένως ε, στο εξωτερικό τι σημαίνει μία τράπεζα με 7% του εθνικού ΑΕΠ. Πρόκειται για μία τεράστια στρατηγική και χρειάζεται απίστευτο τόλμη για να γίνουν αυτά τα βήματα. Κάτι άλλο, ένας άλλος τομέας, ο, το αέριο. Εδώ ασφαλώς το βάρος πέφτει πάνω στον κόσμο, στο λαό της Ουκρανίας. Από την άλλη, οδηγεί και σε μια κατάσταση όπου η Ναύτογκας, η οποία στο παρελθόν εκπροσωπούσε ένα μεγάλο τμήμα του εθνικού χρέους σε διπλάσιους αριθμούς, πλέον σημειώνει ένα μικρό κέρδος. Ελάχιστο, αλλά κέρδος. Τι γίνεται τώρα σε ό,τι αφορά με τον κόσμο, οι τροχονόμοι αν μιλήσει κανείς ε, στον κόσμο, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πλέον δεν σταματάει η τροχέα για δωροδοκίες. Ένας άλλος ε, κλάδος είναι η υγειονομική περίθαλψη και οι συμβάσει στον τομέα της υγείας. Και εκεί δεν υπάρχουν ε, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, διακόπτη ο πρόεδρο. Έχουμε μια άλλη συνεδρία στι 8.30 και έχουμε άλλο ένα σημείο. Δυστυχώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα που μα λέτε, αλλά θα πρέπει να βιαστείτε λίγο παραπάνω. Ναι, όχι, θα σταματήσω στο σημείο αυτό, γιατί νομίζω ότι στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έχουν συμβεί πάρα πολλά και αυτό καθιστά το κράτο πιο διαφανέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φάζακα. Ευχαριστώ, πρόεδρε και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτέ για τα όσα είπατε και όσα ρωτήσατε. Πρώτα-πρώτα θα περιοριστώ αντίστοιχο με τον κύριο Βάγνερ, ο οποίος έχει εντολή να σας ε, ενημερώσει. Εγώ πρέπει να περιοριστώ στα όσα περιέχονται σε αυτήν την έκθεση που ολοκληρώθηκε το 2015. Ο κ. σας είπε τα πιο πρόσφατα. Καλά, άμα θέλετε πάμε σε, για, ένα καφεδάκι και να σας πω τη γνώμη μου για αυτό που ρωτήσατε κυρία Χαουταλά. Αλλά κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένο εκ του ρόλου μου να σας μιλήσω μόνο επί της εκθέσεως. Το θέμα είναι πολύ λεπτό. Ως Ούγγρος ενδιαφέρομαι πάρα πολύ και παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Ουγγαρία. Έχω άποψη από αυτού, αλλά υποχρεώμαι να μην τοποθετηθώ πλευράς πολιτικής ούτε να βγω από τα χωράφια αυτής της έκθεσης. Οπότε ευχαριστώ που φέρατε το θέμα της ε, διαφθοράς. Έχουμε διάφορες προτάσεις εδώ και λέμε ότι Όσον αφορά τα, τη διαχείριση των δημοσιονομικών, αυτό είναι μία από τις προποθέσει για να δοθεί και άλλη βοήθεια και είχε γίνει από ένα χρόνο στην ε, Ουκρανία μία αποστολή και αυτό είναι πέραν τη έκθεση. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο να διαπιστώνει κανείς το πόσοι φορεί πόσοι θεσμοί καινούργοι υπάρχουν κατά τη διαφθοράς στη χώρα. Αλλά εσείς περιμένετε κάποια στοιχεία όσον αφορά την διαφθορά στα ανώτατα επίπεδα. Άρα, ε, για να προχωρήσει η οικονομική αρρωγή, αυτές είναι προϋποθέσεις. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο χρήματος, είναι και θέμα πολιτικής ε, επιρροής. Και αυτός είναι ο του κυρίου Βάγνερ Γίνεται τώρα διάλογος με τις αρχές της χώρας και πάντοτε θα πρέπει να τους τονίζετε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα πρέπει μόνο να ανακοινώνονται, αλλά θα πρέπει και να υλοποιούνται όπως προβλέπετε. Τώρα, όσον αφορά την συνθήκη, δεν ήταν και ούτε αυτό περιεχόμενο τη έκθεση, να σα πω, αλλά τέλο πάντων δεν, δεν ήταν στην εντολή μα. Όσον αφορά την ατιμόγλευση αλλά και την συνεργασία με το διεθνή θεσμικά όργανα στην έκθεσή μα, θα δείτε ότι θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετική, στενή συνεργασία με το Δούνο του και την Παγκοσμία Τράπεζα και είπαμε ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα πρέπει να έχει αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όποιο είναι ο μάστος τη Ορχήστρα, αυτό είναι που πληρώνει. Οπότε πολλές φορές στο Διεθνές Νομισματοταμείο και μια Τράπεζα προτείνουν ότι πρέπει να γίνει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ε, χρηματοδοτούν το, το, το, τα αυτά που δίνονται. Άρα χρειάζεται συνεργασία. Ήταν η συνεργασία στενή και ανέκαθεν το θέμα ήταν οριζόντιο. Ποιο η καταπολέμηση της διαφθοράς Οπότε γι' αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει πρώτα πρώτα να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαφθορά. Αν υπάρχει διαφθορά θα μπει φρένο στις εκταμιεύσεις. Τόσο όλο το θέμα του γενικού εισαγγελέα, αυτό το οποίο έγινε πέρσι, πέρσι και δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση, αλλά ξέρω όλη την ιστορία. Ένα σωρό φορείς συγκροτήθηκαν, αλλά δυστυχώς ακόμα περιμένουμε να ακούσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα αυτών των φορέων σαν αφορά τώρα τη δήλωση, είναι πολιτικό το θέμα. Είναι εκτό θέματο όσον με την αποστολή μα. Ε, και εσεί τα είπατε σωστά πάντω, κυρία Τσέλερ. Τσάιλ. Ε, τώρα όσον αφορά αυτές τις προκαταβολές, αυτού του είδου τα, τα κατεπήγοντα, τα είδα για την αποστολή σας, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να συμμετάσχω γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις. Όμως με χαρά είδα ότι κάνατε ε, κάποιες επικρίσεις όπως και σε άλλες περιπτώσεις και λάβατε υπόψη όμως τη συνθήκες της χώρας ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να συνεχιστούν στο μέλλον αλλά ότι καταρχήν αυτές οι προκαταβολές έχουν τα χαρακτήρα γιατί θα πρέπει κάποια πράγματα να περισσωθούν. αυτά θα απαντούσα εγώ. Αλλά να ευχαριστήσω και τον κύριο Βάγνερ για την ενημέρωση. Μα είπε τις πιο πρόσφατε εξελίξει. και όπως είπα στο συμπέρασμα της έκθεσής μου η βοήθεια την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν. Ήταν πολύ χρήσιμη. Και όπως είπε και ο κύριο Τσέλερ ο εισηγητή, πρέπει να τεθούν κάποιε προποθέσει. Και έτσι να πετύχουν τα αποτελέσματα τα θετικά που θέλουμε για τη χώρα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Φαζέκας για τις ε, απαντήσεις. Όπως πάντα τα είπατε πολύ α, ελαφυρά και είπαμε ότι όπου χρειάζεται πάτε για καφεδάκι και να τα πείτε με τους συναδέλφους. Κύριε Τζέλερ. Ευχαριστώ πολύ, Ερικ. Ε, Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά κατά τα άλλα, Βεβαίως ε, μπορώ να πω ότι έχει απολύτως δίκιο ο κύριος ε, Φάσακας. Ισχύει για την Ουκρανία κάτι που ισχύει και για άλλες ε, χώρες. Η εμπιστοσύνη είναι καλή, αλλά ο έλεγχος είναι καλύτερος. Και αν δούμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ουκρανία, ένα αποτέλεσμα του ταξιδιού μας ήταν ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, δηλαδή σε χαμηλό επίπεδο, επιθυμούν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά στα ανώτερα κλιμάκια υπάρχουν πολλές αντιστάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους νέους αυτούς ανθρώπους να επέλθουν οι αλλαγές στην Ουκρανία. Ε, στο Υπουργείο Εμπορίου είχαμε κάποιες ε, συναντήσεις και μας είπαν ότι οι αποδοχές ε, των ε, στελεχών εκεί είναι εξαιρετικά χαμηλές, ενώ στο ιδιωτικό τομέα είναι πολύ καλύτερες. Όταν ο επικεφαλής της νέας υπηρεσίας για την πάταξη διαφθοράς που συστάθηκε το 2014 μας είπε ότι στο σχέδιο προπολογισμού 2016 το οποίο ψήφισε η Βουλή της Ουκρανίας ε, δεν είχε την ε, δυνατότητα να περάσει η πρόβλεψη κάποιων κονδυλίων για την ε, εκτέλεση εκπλήρωση της δικής του εργασίας, προσωπικό κλπ. Άρα λοιπόν ε, και χρειάστηκε τότε μια παρέμβαση στον ίδιο τον ε, πρόεδρο, ούτω ώστε να τροποποιηθεί το σχέδιο του προπολογισμού. Και αυτός ο επικεφαλής της υπηρεσίας για την πάταξη της διαφθοράς μας είπε ότι αυτόματα χιλιάδες περιπτώσεων που μέχρι στιγμής ε, δεν τις είχαν επεξεργαστεί ήλθαν στο τραπέζι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να διεκπαιρεθούν οι υποθέσεις αυτές από τα παρελθόν γιατί είναι χιλιάδες. Ε, μπορούν μόνο να ασχοληθούν με τις ε, νεότερες υποθέσεις που εφορούν την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ε, χρημάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, κάποιες ε, θετικές ε, προσπάθειες των ανθρώπων που θέλουν να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την κατάσταση της χώρας τους και αυτοί αξίζουν πραγματικά την απόλυτη, την αμέριστη συμπαράστασή μας και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η Πρόεδρος να τους στηρίξουμε όχι μόνο στο Λέμπερκ αλλά και στην Οδυσσό και στο Νεβοπετρόσκα επί παραδείγματι όπου θεωρώ ότι μια τέτοια αρρωγή έχει περισσότερο νόημα ένας ε, επιχειρηματίας ο οποίος ε, έχει μια επιχείρηση αερίου με 117 υπαλλήλους ε, τον ρωτήσαμε και κάνει και εξαγωγές, τον ρωτήσαμε τι προτάσεις, τι συστάσεις θέλει να μας ε, κάνει και μας είπε μη δώσετε καθόλου χρήματα στην ε, κυβέρνηση. Αυτό βεβαίως ήταν μια αγροθιά στο στομάχι. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα εξής. Υπάρχει μια περιοχή όπου υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά δάση και εκεί γίνεται παράνομη υλοτόμηση. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιες εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ο κανονισμός για την εμπορία ξυλίας δεν εφαρμόζεται σωστά από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να παλέψουμε συγχρόνως σε δύο μέτωπα. Ε, κατά τα άλλα χαίρομαι για την ε, περαιτέρω συζήτηση και επαναλαμβάνω ε, υπό το πνεύμα της ενίσχυσης των πολιτών της Ικρανίας θα πρέπει να συνεχίσουμε αλλά θα πρέπει να είναι ορατό ότι γίνεται από τη δική μας πλευρά μεν η προσπάθεια αυτή αλλά θα πρέπει να τελεσφορήσει και να έχει ορατά αποτελέσματα. Να είναι αποδοτική αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δυστυχώς ε, έχουμε ελάχιστο χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο ε, θα έπρεπε να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο. Τώρα θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, η επόμενη συνάντηση είναι στις 8.30 στο κτίριο ΒΙΚ. Ε, δεν έχουμε ελικόπτερο για να πάμε εκεί, άρα μας μένουν 15 ε, λεπτά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. τώρα, το επόμενο σημείο και πάλι συγητής είναι ο κύριος Τσέλερ για την προενταξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και το μεταέλεγχο. Ε, συγγνώμη κύριε Φάσακα, εσείς έχετε πρώτο στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αδύνατη η αποστολή να σας ε, παρουσιάσω αυτή την εξαιρετικά σημαντική έκθεση για τα Δυτικά Βαλκάνια Ε, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν και ο κύριος Τσέλερ και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω. Ε, ίσως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο και όσοι θέλουν να πάνε στις συνεδρίες του ΕΚΟΦΗΝ να φύγουν. Δεν ξέρω. Όχι, πρόεδρος, θα το κάνουμε πολύ σύντομα εάν το αναβάλουμε θα γίνει μετά την απαλλαγή. Δεν ξέρω, κύριο Στσέλλερ, εγώ θα ήμουν υπέρ του να αναβληθεί η συζήτηση. Γιατί θεωρώ επίσης ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, είναι ακόμα πιο εκτεταμένη από την έκθεση για την Ουκρανία και αφορά και περισσότερες χώρες και είναι η πρώτη φορά που το ελεγκτικό συνέδριο έχει διενεργήσει ένα τέτοιο είδους μεταέλεγχο και νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει και τη συζήτηση για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Άρα η πρότασή μου είναι να αναβληθεί. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι λογικό. Άρα λοιπόν συμφωνούμε να αναβληθεί το σημείο αυτό για τον Απρίλιο που θα έχουμε μια πιο δεξιόδικη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Φάτσακας για την πρότασή σας. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ε, συνάδελφοι, θα πράσουμε τώρα στα διάφορα, προσεχείς συνεδριάσεις. To Να στα όσα είπε η κυρία Γκρέσλε, ότι λυπάται που η συμμετοχή σας ε, στην αποστολή στην Ουκρανία δεν περιλάμβανε πολλά μέλη και εγώ της είπα ότι λυπήθηκα πάρα πολύ που είχα προσκληθεί σε αυτή την αποστολή αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Είναι για μένα μεγάλη τιμή κάθε φορά που με προσκαλείτε. Είχα πάει στο παρελθόν δύο φορές στο Βελιγράδι. Αυτή τη φορά ε, το πρόγραμμα αυτό το οποίο επισκεφτήκατε δεν είχε ελεγχθεί από μας. Αλλά δέχομαι την κριτική σας και θα ήθελα να σας πω ότι στο εξής όταν καλείτε τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου να συμμετάσχουν στις αποστολές σας πραγματικά θα δώσουν μια προτεραιότητα σε αυτό και θα ικανοποιήσουν το αίτημά σας. Okay. One final thing. I understand. Ένα τελευταίο σημείο, επιτρέψτε μου, κατανοώ. Ποιος? Ο, ο Διευθυντής ήταν εδώ για να ανοίξει το θέμα αυτό, να μιλήσει εισαγωγικά. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναβολή του θέματος. Και... Ζητούμε συγγνώμη λοιπόν που χρειάζεστε, χρειάζεται να ταξιδέψετε πάλι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε αν υπάρχει κακή οργάνωση στις ε, συνεδριάσεις του Στρασβούργου. Συγγνώμη